από την ευρία αντιπροσώπευση των ενδιαφερομένων. Εγώ προσδοκώ ότι η εθνικότητα επίσης των διευθυντών ε, θα επηρεάσει τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τις ανώτερες θέσεις και να την παρακολουθούμε διότι συμφέρει ολόκληρη την Ένωση η διαδικασία αυτή να υπάρξει διαφανής χωρίς ε, υποψίες προστατευτισμού εντός της ενιαίας αγοράς. Η δημιουργία του ίδιου του οργανισμού της ίδιας της αρχής η διαδικασία η δημιουργίας της είναι κρίσιμη για ολόκληρη την Ευρώπη και για το μέλλον της αγοράς μας. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κύριε Μαριά, για να κλείσουμε αυτό το κατσιδιάι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να στηρίξει την προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ελάχιστου μισθού, αντί να θεσμοθετήσει ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο επίδομα ανεργίας, αντί να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη με κλασική περίπτωση την παραβίαση 1999 της οδηγίας η οποία αφορά τις άτυπες εργασιακές σχέσεις αντί να σταματήσει την ομοιρία χιλιάδων εκπαιδευτικών αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών στην ελλάδα ωρεοποιεί την κατάσταση και μας λέει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αρχή για τα θέματα της εργασίας. πρόκειται για ένα νέο γραφειοκρατικό μηχανισμό μια προσπάθεια υφαρπαγής αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. ας κοιτάξει η ευρωπαϊκή ένωση τις παραβιάσεις που γίνονται καθημερινά και εκεί να δώσει τη δικιά της ενέργεια. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Τάισεν, λόγω σε εσά είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, αλλά σα παρακαλώ να πάρετε το λόγο για να κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Όπω είπα προηγουμένω, η πρότασή μα για τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία υπήρξε το τελευταίο νομοθέτημα της ε, μεταρρύθμισης που ξεκινήσαμε για τη διασφάλιση της ε, ισότιμη κινητικότητα των εργαζομένων. Όταν έλαβα το χαρτοφυλάκιο μου για την απασχόληση, τι ε, κοινωνικέ δεξιότητε και την κινητικότητα των εργαζομένων, ήξερα ότι η κινητικότητα δεν θα ήταν και το ευκολότερο θέμα. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενη που μετά από την αναθεώρηση τη οδηγία για την αποσπάση των εργαζομένων, τώρα σα ζητάμε να ψηφίσετε αυτό τον κανονισμό. Άλλο ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση τη δίκαιης κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη. Υλοποιεί την αρχή του, κοινωνα... του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων σε διασυνοριακό πλαίσιο. Δυστυχώ, δεν έχει καταστεί ακόμα ε, δυνατό για τους συνομοθέτες να συμφωνήσουν στην προτινόμενο εξυγχρονισμό ε, των ε, κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, με βέβαιη ότι η θέση που θα υιοθετήσετε την Πέμπτη σε πρώτη ανάγνωση θα στρώσει το έδαφος για μια επικοδομητική και γρήγορη ελπίζουμε υιοθέτηση μετά από τις ευρωεκλογέ. Τα εκατομμύρια πολιτών για τους οποίους η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί πραγματικότητα καθημερινή ευκαιρία ή μερικές φορές απόλυτη ανάγκη αξίζουν επικαιροποιημένους κανόνες το συντομότερο δυνατόν. Η ελεύθερη κυκλοφορία, αγαπητά μέλη, η ελεύθερη κυκλοφορία υπήρξε θεμέλιος λήθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει να το αποτελεί σήμερα. Ακόμη περισσότερα οι οικονομίες και οι αγορές εργασίας των κρατών μελών μας έχουν, ε, είναι πλέον όλα ένα και πιο συνδεδεμένες και η ελεύθερη κυκλοφορία δίνει ε, τις συνδέσεις μεταξύ των πολιτών μας, των λαών μας. Η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ίση και δίκαιη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Από, όλα αυτά αποτελούν τις αρχές που με καθοδήγησαν στις προτάσεις μας για την ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Αρχές, κατευθυντήριες που μας βοηθούν να οδηγηθούμε σε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα υποστηριχθούν από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά λάβαμε υπόψη σε αυτόν τον κανονισμό για την σύσταση τη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία. Και σα καλώ να την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, κύριε Λενάρτ, παρακαλώ να κλείσετε σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δείχνει πόσο σημαντική είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία στο γεγονό ότι τόσο πολλοί συνάδελφοι ήρθαν στο ημικύκλιο για να μην χάσουν το τέλος της συζήτησης για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Για όσους ήσασταν εδώ από την αρχή, θα ήθελα να πω το εξή. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, πραγματικά. Ιδρύουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, κρίσιμο, προς την ολοκλήρωση μιας πραγματικά δίκαιης και κοινωνικής αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Μέχρι τώρα είχαμε τη, απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Τώρα εξασφαλίζουμε τη δίκαιη κινητικότητα. Μια αγορά εργασίας όπου είναι εγγυημένα και προστατεύονται τα δικαιώματα ε, των ε, εργαζομένων που δεν χωρούν ψευδό αυτοαπασχολούμενοι, κοινωνικό ντάμπινγκ και αθέμητος ανταγωνισμός. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιβάλλονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες και να εφαρμόζονται στον κλάδο της κινητικότητας κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτό είναι ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία και πολύ σύντομα θα αρχίζει να τον υλοποιεί. Είναι πραγματικά ορόσημο και δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει αποτελέσματα σε ένα κλάδο που ε, ανησυχεί και προβληματίζει τους πολίτες και μάλιστα γρήγορα. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επίτροπο την κυρία Τάισεν, τη Ρουμανική Προεδρία και όλους τους συναδέλφους που συνεργαστήκαμε με τρόπο πάρα πολύ ε, αποτελεσματικό και επικοδομητικό για να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Υπολογίζω σε εσά και προβλέπω σε εσά για να επιτύχει στο μέλλον αυτή η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή. Σα ευχαριστώ όλου για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Τελειώνει εδώ η συζήτηση και η ε, ψηφοφορία θα ακολουθήσει σε λίγο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πριν αρχίσουμε τις ψηφοφορίες, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια καλωσορίσουμε την Γκρέτα Τούνμπερκ. Σήμερα έχουμε ενώπιον μας μια εκλεκτή προσκεκλημένη στο θεωρείο των επισκεπτών. Σχεδόν δεν χρειάζεται συστάσεις. Πρόκειται για μια νέα Ευρωπαία πολίτη από τη Σουηδία που με την προσωπική της ιστορία, το σθένος, το θάρρος, τις ιδέες και τη αφήνειά της έχει γίνει σύμβολο της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής ε, λόγω του επίγοντος χαρακτήρα και της μεγάλης σημασίας και φιλοδοξίας του εγχειρήματος. Η Γκρέτα Τούνμπερκ μας πιέζει σε εμά που νομοθετούμε, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να εντείνουμε τις προσπάθειές μας απέναντι στην ε, κλιματική κρίση. Το Μητρό και η ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε αυτή τη θητεία έχει αποδείξει ότι κατανοούμε πόσο φιλόδοξο ε, είναι αυτό το εγχείρημα και συμμεριζόμαστε και τη δική της φιλοδοξία. Μπορούμε να κάνουμε ένα απολογισμό τη θητεία, ξέροντας ότι ανεπιστρεπτή έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο για την προστασία ε, του κλίματος και του περιβάλλοντος. Αν δούμε τι γίνεται με τις εκπομπές των μεταφορών ή με την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών ρήπων. Το Κοινοβούλιο ήταν εκείνο το θεσμικό όργανο που ε, έβαζε πιο ψηλά τον πύχη για να μην αναφέρω την έγκριση και κύρωση ρεκόρ ε, της Συμφωνίας των Παρισιών για την οποία πιέσαμε και την οποία πανηγυρίσαμε παρουσία του τότε Γενικού Γραμματέα ε, του ΟΗΕ Μπαν Κιμούν. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν αρκούν όλα αυτά, ότι θα πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας κάτι σε προσωπικό επίπεδο, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Αν θέλουμε να αποφύγουμε υπερθέρμανση του πλανήτη άνω των, ε, το 1,5 βαθμού Κελσίου και να αποφύγουμε και τη σχετική απερίμωση που ακολουθεί. Η επόμενη θητεία θα είναι κομβική προς την κατεύθυνση αυτή. Η κυρία ε, Τούνμπερκ θα ε, μιλήσει και θα ανταλλάξει απόψη στην Επιτροπή NV στις 2 ε, σε μια συνεδρίαση ανοιχτή σε όλους τους βουλευτές. Σας καλωσορίσαμε ήδη με ένα θερμό χειροκρότημα. Δεν πειράζει, μπορούμε και να το επαναλάβουμε. Καλώς όρισες, Γκρέτα. Oh. Oh. Ε, ε, Ο κύριος Προύστ ζήτησε το λόγο. Euh, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χτες με σφιγμένη την καρδιά, οι Καθολικοί, οι Παριζιάνοι και οι Γάλλοι είδαν ε, την Παναγία των Παρισίων στις πλόγες. Θέλω εδώ λοιπόν να εκφραστώ εκ μέρους της γαλλικής αντιπροσωπείας και είμαι βέβαιος και εκ μέρους όλων σας την βαθιά μας θλίψη απέναντι σε αυτή την καταστροφή. Πρόκειται για ένα θησαυρό της, του γαλλικού πολιτισμού που καταστράφηκε εν μέρη. Ε, ε, έπιασε φωτιά ένα γλυπτό του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με αυτό κάηκε και η καρδιά μας. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν όλη τη νύχτα ε, την πυρκαγιά για να μείνει όρθια η Εκκλησία. Σας το λέω, η Γαλλία και οι Γάλλοι θα παραμείνουν σταθεροί, θα έχουν αντοχή απέναντι σε αυτό το γεγονός. Θα την οικοδομήσουμε και πάλι αύριο. Θέλω αγαπητοί συνάδελφοι να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας προς τη Γαλλία. Σε αυτό το θησαυρό της εθνικής μας κληρονομιάς και για τον οποίο φροντίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Όπως έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό στην Παναγία των Παρισίων, κάθε άνθρωπος, κάθε άτομο προσφέρει το λιθαράκι του και εμείς θα προσφέρουμε το δικό μας για την ανοικοδόμηση αυτού του συμβόλου. Σας ευχαριστώ. Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι που θα κρατήσει ένα δευτερόλεπτο. Το 1963, ε, όταν ξεκίνησε η κατασκευή, υπήρξε ειδική, υπήρχαν ειδικοί εργαζόμενοι για την, την ε, λιθογλύπτες όχι μόνο από τη Γαλλία, αλλά από όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμα και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που ήρθαν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση αυτού του μνημείου του πολιτισμού. Δεν ήθελα όμως να πω αυτό. Κύριε Πρόεδρε, με ονομάσατε ε, πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας σε αυτήν την ε, θητεία μαζί με άλλους συναδέλφους. Στη διάρκεια αυτής της θητείας Υποστήκαμε πολλές πιέσεις από λόμπι τα οποία εγκαταστάθηκαν στο ε, Κοινοβούλιο. Θέλω να σας υπενθυμίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι κατά την ψήφιση των, ε, για την οδηγία των δικαιωμάτων του δημιουργού υπάρχουν λομπίστες. Και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον όσον και την διαθεσμική φάση. Θα ήθελα να αφήσετε την, στο επόμενο κοινοβούλιο την υποχρέωση να ενισχυθούν οι κανόνες που εμποδίζουν το λόμπι από τη στιγμή που ένα κείμενο φτάνει στην Ολομέλεια ε, και αυτό να περάσει στο επόμενο κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθούν οι ψηφοφορίες. Πρώτη έκθεση. Έκθεση Βίξτρομ. Κοινοτικέ στρατι... στατιστικέ για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με 492 ψήφους υπέρ, 109 κατά και 35 εποχές. Το Κοινοβούλιο ολοκληρώνει ούτω την πρώτη του ανάγνωση. Δεύτερη έκθεση Τη κυρία Γοζιέχ. Αλλά ζητεί το λόγο η κυρία Τέισεν πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Κομισιόν στηρίζει τη σύσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, συν, να ε, προσχωρήσει στην πράξη της Γενέβης. Παρ' όλα αυτά, η θέση της Κομισιόν διαφέρει από τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου όσον αφορά την δυνατότητα όλων των κρατών μελών να ενταχθούν στην πράξη της Γενέβης λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επ' αυτού. Κατ' εξαίρεση, θα μπορούσε να συμφωνήσει η Κομισιόν στην συγκεκριμένη περίπτωση τα επτά κράτη-μέλη που έχουν συνυπογράψει τη Συμφωνία της Λισαβόνας ε, επί πολύ καιρό θα μπορούσαν να ε, προσχωρήσουν στην πράξη της Γενέβης εκ μέρους της Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στη δήλωση της Κομισιόν η οποία έγινε σχετικά και η οποία υποβλήθηκε και στο Συμβούλιο και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμα μέλη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τάισεν και προχωρούμε στην ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Εγκρίνεται η έκθεση. Άλλη έκθεση Γοζιέρ. Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική. Σε Πέρας. Εγκρίνεται. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ψήφι είναι δυνατά σου χειρός αυτή. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το κοινοβούλιο ολοκληρώνει την πρώτη του ανάγνωση. Έκθεση Ράντος. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Σε la Εγκρίνεται. Έκθεση Φορέντζα. Με ονομαστική κρίση. Α, θέλει το λόγο η συγγήτρια. Παρακαλώ για δύο λεπτά, κύριε Φορέντζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα αυτή τη σύσταση, διότι η παραγωγή ελαιολάδου είναι σημαντικότατο τομέα για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, για την οικονομία των μεσογειακών χωρών, για την Ιταλία ε, η ποιότητα των προϊόντων έχει πληγεί από, διάφορες, ε, από διάφορους επιβλεβείς οργανισμούς, ε, από την παγωνιά. Οπότε θέλω να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στη διεθνή συνεργασία για την παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπεζών ελαιών. Ωστόσο, λυπάμαι για την καθυστέρηση με την οποία διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η συμφωνία και η έλλειψη πληροφοριών, έγκυρων πληροφοριών από τα άλλα θεσμικά όργανα για τι διαπραγματεύσει. Οι συμφωνίε που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν τη συνένεση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο, καλό το Συμβούλιο και την Κομισιόν να ενημερώνουν επαρκώ το Κοινοβούλιο ειδικότερα όσον αφορά οποιαδήποτε απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί σε σχέση με το άρθρο 4 της απόφασης του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. Με στην κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Τάραντ. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Δύο λεπτά το πολύ, παρακαλώ, κύριε Τάραντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρω πως δεν μας αρέσουν οι ομιλίες των εισηγητών που διακόπτουν την ομαλή ροή των ψηφοφοριών. Δυστυχώς όμως σήμερα είμαι υποχρεωμένος να εξηγήσω τα διλήμματα που έχουμε ενώπιόν μας. Όλοι γνωρίζουμε πόσες φορές γελάει ο αστυνομικός όταν του λες αστείο. Όμως στη θητεία αυτή είχαμε οκτώ διορισμούς στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και με την εξαίρεση τη Ιρλανδίας ήταν πολιτικές. Και πρέπει να πω ότι όλο και περισσότερο από τα νεότερα ε, κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων η Ιστονία, η Φιλανδία και η Ουγγαρία. Δεν λέω ότι οι πολιτικοί είναι ακατάλληλοι ή ανίκανοι να κάνουν κάποια άλλη επαγγελματική εργασία. Αντίθετα η κυρία ε, έχει πολύ καλή βιογραφία γραφικό. Όμως οι διαδικασίε επιλογής των υποψηφίων τα κράτη-μέλη δεν είναι διαφανεί. Στρέφομαι προς τα κράτη-μέλη και του ζητώ να ακούσουν την κλίση του Κοινοβουλίου και πάντοτε να, να υποβάλουν δύο υποψηφίους και να ακολουθήσουν το ε, ε, ε, το παράδειγμα της Ιρλανδίας δηλαδή να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός υπό το πνεύμα του άρθρου 255 ε, των συνθήκων. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σκεφτούμε αν χρειαζόμαστε ταυτόχρονα μέλος του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου εκ μέρους όλων των κρατών μελών. Γιατί να έχουμε 14 ελεγκτές στη μία περίοδο και 14 στην άλλη. Αν, αποτύχουμε θα είναι λιγότεροι, θα είναι περισσότεροι απογοητευμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, ψηφίστε όπως προτείνει ο εισηγητής αυτή τη φορά, αλλά μην ξεχνάτε ότι η διαδικασία των κυβερνήσεων Ρουμανίας και Κροατίας δεν ήταν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σύμφωνα με την τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελικά ο, ο, ο αστυνόμος μια φορά μόνο γελάει όταν του λες αστεία. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. Μυστική ψηφοφορία. Cerramos la votación. Απορρίπτεται. Informe Tarant, propuesta... Άλλη έκθεση Τάραντ, προτινόμενος διορισμός μέρους του ελεκτικού συνεδρίου. Sí. Θα ήθελα να θυμίσω στον συνάδελφό μου ότι σήμερα ψηφίζουμε ε, σύμφωνα με τη συνήθεια διαδικασία και ήταν πολύ ιδεολογική ε, ομιλία αυτή που ακούσαμε, που κανονικά δεν θα πρέπει να την ακούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποφασίστε με κριτήρια αξιοκρατικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πάλι μυστική για το διορισμό της κυρίας Ιβάνα Μάλετιτς. Σε ψηφοφορία. Πέρας Αγκρίνεται. Έκθεση Ροζιέ. Η προσωρινή συμφωνία 155. Η τροπολογία έρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 156, δήλωση της Επιτροπής Δυνατάς Χειρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώνει έτσι την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβούλιο. Έκθεση κλίντς με ονομαστική ε, κλίση αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας, ορίστε. Ο εισηγητής ζήτησε το λόγο. Εγκρίνεται. Μπορώ να έχω το λόγο, λέει ο κύριος Κλίντς. Παρακαλώ. Σύντομα, σύντομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 15 χρόνια θα αποχωρήσω από το Κοινοβούλιο στο τέλος της αιτία μου. Έχω τις δύο τελευταίες μου εκθέσεις σήμερα και μου έδειξε η εργασία μου για τι εκθέσει αυτέ ότι το Κοινοβούλιο μπορεί και γέφυρε να χτίσει και συνένεση να βρει σε ε, αντίθεση με πολλά εθνικά κοινοβούλια. Πολλοί από εσά θα είστε και πάλι υποψήφοι και θα εκλεγείτε ευρωβουλευτές. Θέλω να απευθύνω έκκληση προς όλους σας να μην χαλαρώσετε τον αγώνα υπέρ των ευρωπαϊκών ιδεοδών. Πάνω από 60 χρόνια μα έχει εξασφαλίσει κράτος δικαίου, δημοκρατία, ελευθερία, δικαιώματα και σχετική εφημερία. Το οφείλουμε στα παιδιά μα και ε, στα εγγόνια μας να μην αποτύχει το ευρωπαϊκό ε, εγχείρημα και να παραμείνει ε, η η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι το μοναδικό μας μέλλον, δεν έχουμε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σεγετά. Ολοκληρώνει λοιπόν την πρώτη ανάγνωσή του το Κοινοβούλιο. Δεύτερη έκθεση κλίντς με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Και τελειώνει. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση Σίμων με ονομαστική ε, κλίση, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Και άλλη έκθεση Σίμων, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνει έτσι το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Έκθεση Χιόκμαρκ. Με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Α, κύριε Χιόκμαρκ, έχετε το λόγο. Um, ε, όπως και ο κύριος Κλίμπ, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καταπληκτικά αυτά 15 χρόνια, για τους εξαιρετικούς φίλους από όλους τους χώρους ε, πολιτικούς και γεωγραφικούς και θέλω να πω ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πιο ισχυρή την Ευρώπη, μια ελεύθερη κοινωνία ανοιχτή σε όλους, δυνατή σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χρειάζεται συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το γοητευτικό, εντυπωσιακό. Πολλές φορές έχουμε διστάμενες απόψεις, αλλά σημασία έχει ότι έχουμε κοινό καθήκον και κοινό στόχο. Σας ευχαριστώ όλους για τα καταπληκτικά αυτά 15 χρόνια. Πρόκειται για τις δύο τελευταίες μου εκθέσεις που ελπίζω θα βοηθήσουν στη σταθερότητα της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρα. cierra la votación. Aprobado. Εγκρίνεται. Και ολοκληρώνει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Δεύτερη έκθεση Χιόκμακ. Αρχίζει και πάλι η ψηφοφορία ονομαστικά. Πέρας. Aprobado. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνει έτσι το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Έκθεση Φερνάντε. Πρώτη τροπολογία. Δυνατά σου χειρό Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται ακριώνει το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Έκθεση κάρα και μπερέ. Τροπολόγια 2 με ονομαστική κλίση αρχή ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Κυρία Μπερέ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περίμενα την ψήφο της τρίτης έκθεσης. Όπως οι συναδελφοί Βολφ Κλίντς και Χοκμαρ, ε, μόνο μετά από 25 χρόνια, μόλις μετά από 25 χρόνια αυτή θα είναι η τελευταία μου έκθεση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, όσοι αγωνίστηκαν μαζί μου, με όσους ε, τσακώθηκα ή συμφώνησα με όσους καταλήξαμε να βρούμε μια ευρωπαϊκή θέση. Να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, όλους του υπαλλήλου ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας πω ότι εγκαταλείπω ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έχει αλλάξει ριζικά. Και εμείς οι ίδιοι έχουμε αλλάξει, η Ευρώπη έχει αλλάξει. Αλλά το Κοινοβούλιο αυτό έχει γίνει πλέον ένα πραγματικό Κοινοβούλιο των πολιτών. Πάντα λέμε ότι ακούει υπερβολικά τα λόμπι, αλλά είναι συντονισμένο και με αυτό το κύμα Ευρωπαίων που γίνεται όλο και δυνατότερο και που είναι πεπισμένο ότι η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέλλον για αυτούς. Ε, το κοινοβούλιο αυτό είναι σύγχρονο, γνήσιο, δημοκρατικό, αυθεντικό. Είναι το κοινοβούλιο των πολιτών. Να το κρατήσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπερές. Δεύτερη έκθεση Κάρας Μπερές με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ολοκληρώνεται έτσι λοιπόν η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Και άλλη έκθεση, Κάρας Μπερές, με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνει έτσι το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Έκθεση Φέρμπερ. Με ονομαστική κλίση, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται, ολοκληρώνει το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Άλλη έκθεση Φέρμπερ, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνει το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Έκθεση Καλβέτ Σαμπόν. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Καλβέτ. Α, όχι, δεν το ζήτησε. Η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο προηγουμένως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βάσει του άρθρου 159 εδάφιο 3 του κανονισμού θα ήθελα να ζητήσω ε, ονομαστική διαδικαστική ε, ψηφοφορία για να ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες πριν την προσωρινή συμφωνία. Ε, οι τροπολογίες αυτές έρουν διακριτικές εξαιρέσεις στην εφαρμογή της οδηγίας και έτσι εξασφαλίζουμε προστασία του συνόλου των εργαζομένων, κυρίως εκείνων που ε, βρίσκονται σε επισφαλή θέση, όπως είναι οι οικιακές βοηθοί και η ναυτική. Παρακαλώ λοιπόν διαδικαστικά να ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες. Ε, ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σέβομαι ε, τις εξαιρετικότατες προθέσεις και πιθανότατα συμμερίζομαι και τις απόψεις που κρύβονται πίσω από τις ε, ε, αιτήσει αυτές, γιατί και εγώ το ήθελα, αλλά δεν μπόρεσα να το αποφύγω, αλλά για το καλό της κοινοβουλευτική εργασίας και για το καλό της έκθεσης που περιέχει πολύ περισσότερα από αυτά, σας παρακαλώ για να σεβαστούμε την ισορροπία που ήταν τόσο δύσκολο να επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις, σας παρακαλώ να μην γίνει δεκτό αυτό το αίτημα και να ψηφίσουμε το κείμενο ε, χωρίς να το κάνουμε πιο εύθραυστο. Ε, ευχαριστώ. Θέτω σε ηλεκτρονική ψηφοφορία την πρόταση της κυρίας Λόπεθ Μπερμέχο. Παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη το αίτημα. Οπότε θα ψηφίσουμε κανονικά. Τροπολογία 134 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η δήλωση της Επιτροπής Δυνατά χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνει έτσι το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Κύριε Καλβέτ, θέλετε το λόγο. Τριάντα δεύτερα όμως, παρακαλώ. Με σαμποτάρουν εδώ, Πρόεδρε. Σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία. Είναι το τελευταίο κείμενο σε τούτη εδώ τη θητεία, διότι σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύτος όλο το Κοινοβούλιο, όλους εκείνους που ήταν υπέρ ή κατά, ε, όλη μου την ομάδα, την Ρουμανική Προεδρία και την κυρία Τάισεν, γιατί ε, βάλαμε αυτό το ορόσημο στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκληρωση, της κοινωνικής Ευρώπης, γιατί με πολύ μεγάλη τιμή θα πάρω ως ενθύμιο ε, ε, το κείμενο αυτό από την παρουσία μου εδώ και το πέρασμά μου από το καταπληκτικό αυτό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Ωραία, ψηφίζουμε την έκθεση Λένας. Ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κοινή δήλωση, η τροπολογία 105, δυνατά χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώνει έτσι το Κοινοβούλιο την πρώτη ανάγνωση. Έκθεση Μάτο. Κύριε Μάτο, ζητήσατε το λόγο κι εσείς. Gracias, presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι είχαμε εκατοντάδες συνεδριάσεις, τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, δύο απόπειρες ε, ε, αναθεώρηση αυτού του κανονισμού. 30 κανονισμούς έχουμε συνενώσει και παρακαλώ να υπερψηφιστεί αυτή η συμφωνία που ήταν εύθραυστη, δύσκολη, αλλά που γνώρισε τελικά πολύ μεγάλη συνένεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριος Βαντάλεν, βάση ε, του άρθρου 59, δάφιο 3, θεωρώ ότι είναι απολύτως ε, απαραίτητο να γυρίσει πίσω η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το παράρτημα 5.1 εξ ονόματος των Ολλανδών αλλιέων. Κοιτάξτε τι έχει γίνει εδώ μια τέτοια οικογένεια που εργάζεται με αυτή την ηλεκτρική αλία κινδυνεύει να καταστραφεί στο μέλλον τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Γιατί ακούσαμε για παιδιά και εγγόνια. Στραγγαλίζουμε υπάρξεις τώρα και θέλω να ψηφιστούν χωριστά αυτά και παρακαλώ τους συναδέλφους ε, που υποστηρίζουν το αίτημά μου να αγερθούν αυτή τη στιγμή. Ε, το σκάφος που είναι, γιατί σας βλέπω πολύ εξοπλισμένο, λέει ο Πρόεδρος.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 36, 37, 38. Sí, los hay. Sí. Los hay. Entonces ahora ya votamos. Perfecto. Τρα, Tranquilízase, sí. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ησυχάστε. Έχουμε πάνω από 38. Ωραία. Θα ψηφίσουμε την πρόταση του κυρίου Βαντάλεν, διανατάσσεως χειρό. Ο κύριος Μάτο... Όχι, ο κύριος Ζαντό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εντυπωσιακό που μία από τις ψηφοφορίες που κατέκλυσε την ε, κοινή γνώμη στην Ευρώπη υπέρ των οικοσύστηματων, υπέρ των μικρών αλλιέων κατά της βιομηχανικής αλλίας ήταν τεράστια ε, το θέμα αυτό. Συζητήσαμε γι' αυτό σε όλες τις χώρες και εγώ απαιτώ από αυτό το κοινοβούλιο να διατηρήσει, να κρατήσει την υπόσχεσή του για τα οικοσυστήματα και για τους μικρούς αλληλείς ε, σε όλη την Ευρώπη κατά τη βιομηχάνηση της αλληλείας και κατά της ε, ε, οικονομικής αλληλείας. Ευχαριστώ. Κύριε Μάτο, θα ήθελα μόνο να πω ότι είμαι κατά του αιτήματο του κυρίου Βαντάλεν για τον απλούστατο λόγο αυτό που θέλει με την τροπολογία του είναι να καταργήσει την συμφωνία που είναι τη συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου να τερματιστεί, να απαγορευτεί αυτή η ηλεκτρική αλεία. Αυτή την εντολή έχουμε και αυτή την εντολή ζητώ να υπερψηφίσετε. Άρα να καταψηφίσετε το αίτημα του κυρίου Βαντάλεν αυτή τη στιγμή. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση του κυρίου Βαντάλεν. Διανατάσσου χειρός. Ψήφι κατά αποχές απερίφθη το αίτημα προχωρούμε ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα πέρας εγκρίνεται ολοκληρώνει το κοινοβούλιο έτσι την πρώτη του ανάγνωση έκθεση Λεβαντόφσκι με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση της κυρίας Γκρέσλε. Τροπολογίε 1 έω 4, 7 εω 7, 110, 114, 140. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνονται. Η τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ. ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Πέρασε. Απερίφθη. Η τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 112 ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 142 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Η ψηφοφορία. Για πέρας. Απερίφθη. Οπότε καταπίπτει η επόμενη 141. Ψηφίζουμε ονομαστικά το σύνολο της πρότασης της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση πόσπισιλ. Δυνατός ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση γραπίνη. Δυνατός ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, ε, τροπολογίες 62 και 71. Ε, ονομαστική κλίση τώρα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέρασε. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση Μαμίκενς με ονομαστική κλίση. Είναι η τροπολογία 42. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβούλιο. Το λόγο έχει ο κύριος Μαμίκινς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία των κανονισμών που μόλις εγκρίναμε σήμερα. Είναι ζωτική σημασία γιατί ε, αντιμετωπίζει τις διάφορες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις που γίνονται με αυτοσχέδιες βόμβες και ε, χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες, συμπατριώτες μας θα είχαν σώσει, γλιτώσει τα τελευταία χρόνια αν υπήρχε αυτή η απαγόρευση στους πρόδρομες ουσίες. και πρέπει να ρυθμιστούν ε, οι πωλήσει αυτών των πρόδρομων ουσιών και το κάναμε. Έχουμε ευρία ε, στήριξη αυτού του αποτελέσματος και αυτό φάνηκε στην Επιτροπή. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον όλους τους συναδέρφους για την υποστήριξη στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου, όπως επίσης και για τη μεγάλη συσπήρωση. Ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση Η Τροπολογία 77. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 78. Διανατάσεως ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνει έτσι το κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Έκθεση Λέναρς. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 326. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση μέλο. Η τροπολογία 312 με ονομαστική κλίση αρχής ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση Κιέγγε. Η τροπολογία 69 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Σε la Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση. Το λόγο ζητάει η συγκήτρια. Παρακαλώ, κύριε Κιέγγε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την υιοθέτηση αυτού του κανονισμού κάνουμε άλλο ένα βήμα για την πολιτική διαχείριση της μετανάστευσης. Ευχαριστώ τους και ηγητές. Με υποστήριξαν στεναρά σε αυτή τη διαδρομή. Με μεγάλη αίσθηση ευθύνη ε, βοηθήσαν ε, στην ταχεία υιοθέτηση του κανονισμού. Ελπίζω στην επόμενη θητεία να επανέλθουμε σε αυτό το Κοινοβουλίο να επανέλθω εγώ ώστε να συνεχίσω το έργο μου για αυτό το θέμα με μεγάλη ευθύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη έκθεση και τελευταία είναι της κυρίας Τούν. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, δεν σας αποχαιρετώ. Συνεχίζω να αγωνίζομαι, να αγωνίζομαι για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω να υπερψηφίσετε την έκθεση αυτή που έχουν, υπάρχει ενώπιόν μας. Διότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε ανθρώπους, χιλιάδες Ευρωπαίους από το θάνατο σε τροχαία ατυχήματα. Θα σωθούν πολλές χιλιάδες άνθρωποι από σοβαρούς τραυματισμούς. Το σύστημα αυτό θα προστατεύσει τους πολίτες. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Τα συστήματα αυτά θα εγκατασταθούν στα νέα οχήματα και άρα θα κάνουν ασφαλέστερους τους ευρωπαϊκού δρόμους όχι μόνο για τους οδηγούς και τους επιβάτες τους αλλά κυρίως κυρίως για τους ευάλωτους χρήστες των δρόμων, τους ποδηλάτες, τους πεζούς και άλλους. Και τέλος, η οδική ασφάλεια είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο βοηθά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές μέσω της καλύτερης συνεργασίας, η μεγαλύτερη ασφάλεια, η οδική ασφάλεια είναι χειροπιαστό παράδειγμα ε, για το πώς έχει βελτιωθεί η ασφάλεια στην Ευρώπη και στην καθημερινή μας ζωή. Και όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατανοήσουν απλά και μόνο ότι αφού, την κατάσταση αφού έχουν υποστεί τη ζημιά ζημιά. Είμαστε λοιπόν πολύ περήφανοι και φωνάζουμε για τα επιτεύγματά μας. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 110 με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. δήλωση Επιτροπής 111, τροπολογία δυνατά χειρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώνει έτσι το Κοινοβούλιο την πρώτη του ανάγνωση. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι.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 Κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Το λόγο έχει ο κύριος Μέσεριτς για την έκθεση που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Κύριε Μέσσερσνικ. Είμαι εδώ. Έχουμε μια εσωτερική αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν πιο πλούσιοι και να είναι πιο ασφαλείς. Αλλά δεν τους διασφαλίζει ανάπτυξη και ασφάλεια αν οι χώρες δεν εφαρμόζουν κανόνες ε, σωστά αλλά κερδοσκοπούν ή επινοούν διαφορούς κανόνες ε, που ωφελούν αυτές τις ίδιες εις βάρος των υπολείπων. Εγώ έχω ζήσει την εμπειρία του πώς τα κράτη-μέλη ε, καταφέρουν να υλοποιούν κανόνες ε, μέχρι σήμερα. Πολλά κράτη-μέλη θα έπρεπε να είχαν μάθει πώς να εφαρμόζουν ε, τους κανόνες και ποιοι είναι οι κανόνες, αλλά πάντα υπάρχουν περιπτώσεις χωρών που δεν τους εφαρμόζουν με συνοχή, ενώ αυτή η συνεκτική εφαρμογή είναι απαραίτητη για να έχουμε την ίδια ευημερία παντού. Αλλά και υπό ένα πνεύμα αλληλεγγύης ε, εντός ενίας αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, εγώ αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ και να υποστηρίξω αυτή την οδηγία γιατί έχει ένα σημαντικό σκοπό. Θέλει να προστατεύσει όλους όσοι έχουν αντιληφθεί ότι έχουν υποστεί παραβίαση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και θέλουν να ενημερώνουν για αυτές τις παραβιάσεις. Ε, συμφέρει του λαού μας να γίνεται αυτό και συμφέρει να προστατεύουμε και τους καταγγέλτες δημοσίου συμφέροντό ώστε να μην αποτελούν το αντικείμενο εκβιασμών. Ωστόσο, ε, πρέπει να προσέχουμε τις σημαντικές σύγκρουσεις συμφερόντων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων οι εργοδότες θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες ε, εντό των οποίων οι εργαζομένοι θα μπορούν να καταγγέλνουν παραβιάσεις εργασιών με ασφάλεια. Μην ξεχνάμε επίσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες δεν θέλουμε να περιπλέκουμε τα πράγματα υπερβολικά. Συμφωνώ επίσης με το ότι οι οι εργαζομένοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν εσωτερικέ διαδικασίε πριν καταγγείλουν οτιδήποτε. Ευχαριστώ κύριο Στρογεύσκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα λάβαινα το λόγο σήμερα αν είχα παραστεί στη χθεσινή συζήτηση. Δύο πράγματα με ανησύχησαν. Πρώτον, η έλλειψη σεβασμού για την οδηγία από περιφερειακές δυνάμεις που αυτό που επιδιώκουν είναι να περιπλέξουν τη ζωή των ανθρώπων και να επιτρέψουν τις ε, επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις να είναι υπεράνω του νόμου. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι διαδίδουν ψεύτικες πληροφορίες. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, αλλά έχουμε και μάρτυρες οι οποίοι κακόβουλα, χωρί χωρίς τεκμηρίωση, διαδίδουν φήμες κατά ανθρώπων και επιχειρήσεων και τους καταστρέφουν ψυχικά και ε, οικονομικά. Πρέπει να βρούμε σωστή ε, ισορροπία και αν δεν το κάνουμε θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μορέλ, σε αυτές είναι για την προστασία των προσώπων που καταγγέλουν παραβιάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνέταξε ένα κείμενο πολύ προστατευτικό για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, αλλά το ε, Συμβούλιο το αποδυνάμωσε στη πρέπει να κινητοποιηθούμε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν θα πρέπει να ενημερώνεται ο ανώτερος ιεραρχικά πριν την αποκάλυψη των πληροφοριών. Επίσης, όσοι έχουν ε, συνεισφέρει στην αποκάλυψη αλήθειας θα πρέπει να προστατεύονται. Υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά την αποκάλυψη ε, ε, πληροφοριών, εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την άμυνα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι το πνεύμα, κατά, ας πούμε, σε σχέση με τον Ζουλιάν Σάνζ, όπου περιορίζοντας ε, την, την αρχή αυτή διαφώτσαν την κοινή γνώμη σε, στην περίοδο του πολέμου του Ιράκ. Η ουσία είναι εδώ, το κείμενο είναι καλό και ε, υπάρχει, παρέχει, παρέχει προστασία και άρα ε, κάναμε καλά τη δουλειά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Η παραβίαση του κοινοτικού δικαίου είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι αντιευρωπαϊστές ε, για να δημιουργήσουν θυμό στους ανθρώπους κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πολλοί δεξιοί πολιτικοί προσπαθούν να αποκομίσουν ωφέλη από το γεγονό ότι δεν είναι άριστα σχεδιασμένη η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι όλε οι νομοθεσίε. Όλε οι νομοθεσίε έχουν αδύναμα σημεία και πρέπει να δώσουμε τη μέγιστη ελευθερία στου πολίτε μα να καταγγέλουν τέτοιε αδυναμίε για να συμμετέχει καλύτερα ο, ο κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική. Θα πρέπει να του παρασούμε τα εργαλεία. Εμεί λοιπόν που υπερασπιζόμαστε μια ισχυρή, ολοκληρωμένη Ευρώπη πρέπει να ηγηθούμε τέτοια, ενός τέτοιου αγώνα. Η κακοδιαχείριση εκφράζεται με διάφορους τρόπους, σχέσεις ε, εργασίας, ε, σχέσεις με την ε, σχετίζεται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε περιπτώσεις καταγγελίας πρέπει να παρέχουμε εγγύησεις στους καταγγέλλοντες. Αυτό ήθελα να παρασπίσω, συναδελφοί. Ευχαριστώ. Κύριος Χάναν έρχεται η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι είσαι ένας από τους παλαιότερους στο Κοινοβούλιο. Είμαι αρκετά μεγάλος, θυμάμαι την υπόθεση Τίλακ, όταν ένας γερμανός δημοσιογράφος συνελήφθη επειδή τελικά αποκάλυπτε την απάτη της, της ε, αρχές καταπολέμησης απάτης. Κανένας δεν είχε δει βεβαίως τα προσωπικά χαρτιά. Ή την υπόθεση Μαρκ Αντρίεσιν, όταν ένας λογιστής ήρθε για να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της Κομισιόν και αποκάλυψε ότι σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούσε διπλό εγγραφές και η, υπήρχε μια αντίδραση. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Όλοι οι οργανισμοί ενδιαφέρονται για την αυτοπροστασία του. Αυτό είναι ανθρώπινη φύση, δεν ε, υπάρχει μόνο στις Βρυξέλλες αλλά επιδεινώνεται από την, τον εκφοβισμό ε, και την θρησκευτική πίστη που έχουν πολλοί στο ευρωπαϊκό έργο και που, θεω, του κάνει να θεωρούν ότι η ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αντιμετωπίστε αυτό και θα λύσετε πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ, κυρία Ρούανα. arvoisa puhemies epäkohdista kuten erilaisista rahavarojen ja muun omaisuuden väärinkäytöksistä veronkierrosta ja muista. όσον αφορά tis periptosis apatis φοροδιαφυγής παντός είδους εγκλήματα το ότι κάποιος τα καταγγέλει αποτελεί προϋπόθεση για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν ε, οι καταγγέλτες αυτοί έχουν εμπιστοσύνη ότι θα ε, είναι προστατευμένοι, μπορούν να το κάνουν και έτσι να γίνουν έρευνες κατά ατόμων που θα μπορούσαν να κάνουν τεράστιες ζημιές κατά ατόμων, επιχειρήσεων και κρατών. Ε, και τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Μπορεί να υπάρχουν καταγγέλτες εντός οργανισμών ή απευθείας από τις αρχές. Προστατεύονται από αντίπεινα, από απολύσεις ε, ή από αποκλεισμό. Είμαι ικανοποιημένη που επιτέλους καταφέρνουμε να προστατεύσουμε τέτοιου ανθρώπου με κανόνε, ενώ τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν σχετική νομοθεσία. Η οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί λοιπόν το συντομότερο δυνατόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόλτσακ. Και εγώ